δύο αιτήσει για διορισμό σε αντιπροσωπείες και εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ήδη αυτές οι αιτήσει. Η κυρία Φρουντσούλικα προτείνεται να είναι μέλος της αντιπροσωπείας με την Κορεανική Χερσόνησο και ο Μιχάη Τουρτσάνου ως ε, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και επίσης ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τον Καναδά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επικυρώνονται αυτοί οι διορισμοί.